Dear colleagues, Συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Καθίστε παρακαλώ. Πρόκειται για την κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών ΕΚΟΝ και ΛΥΜΠΕ Έχουμε δύο πάρα πολύ σημαντικά νομοθετικά κείμενα μπροστά μας. Καθίστε παρακαλώ. Επαναλαμβάνω καθίστε. Θα πρέπει να ελέγξουμε το σύστημα ψηφοφορίας και θα πρέπει να δούμε αν έχουμε ε, απαρτία. Όσοι δεν έχουν κάρτες παρακαλώ να μας ενημερώσουν αλλά έτσι και αλλιώς θα πρέπει να κάνουμε μια δοκιμή. Ζητώ από τα μέλη να βάλουν τις κάρτες τους και να ψηφίσουν. Άρχεται η ψηφοφορία, δοκιμαστική ψηφοφορία, δοκιμαστική, άρχεται η ψηφοφορία. Η κυρία Γκόμες ζητάει το λόγο. δεχτήκατε την πρότασή μου, την οποία δεν σας είπα ποια είναι, αλλά τη δεχτήκατε. Υπάρχει απαρτία λοιπόν, τελειώνει η δοκιμαστική ψηφοφορία. Λοιπόν, τώρα μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες. Όπως είπα έχουμε δύο πάρα πολύ σημαντικά έγγραφα. Το πρώτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ήταν και μια μεγάλη επιτυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια του άρθρου 55 η συνεργασία μας ήταν ιδιαίτερος αποτελεσματική των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών. Να συγχαρώ τους Κάρινς και Σαρτζεντίνη, τους εισηγητές και τους Κιώδης για την κατάληξη του τριμερούς ε, διαλόγου για την ομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Όπως επίσης και το θέμα του Μητρώου είναι βασικό επίτευγμα του Κοινοβουλίου. Η διαδικασία τώρα, <clears throat> συγγνώμη, μας οδηγεί στο να ψηφίσουμε την πρώτη ανάγνωση επίσημα του Συμβουλίου. Αλλά βέβαια η πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου είναι αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου. Είναι δηλαδή το κοινό κείμενο στο οποίο έχουμε καταλήξει στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου. Θέτουμε λοιπόν τώρα σε ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία, την πρώτη ανάγνωση, το κείμενο της πρώτης ανάγνωσης του Συμβουλίου για την οδηγία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Άρχεται η ψηφοφορία, ονομαστική, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Δεκτή η πρόταση. Τώρα θα φέσουμε σε ψηφοφορία το κείμενο του Συμβουλίου για τον κανονισμό που αφορά τα συνοδευτικά στοιχεία των μεταφορών χρηματικών ποσών συμπληρωματικό έγγραφο με το προηγούμενο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζεται. Vote is closed. Τέλος της ψηφοφορίας. Δεκτό και το κείμενο αυτό. Συγχαρητήρια στους εισηγητές Κίρκοπ και Σιμών. Ολοκληρώσαμε την διαδικασία. Τέλος της συνεδρίασης. Ε, very long negotiation concluded. How long? Two years. Δύο χρόνια κράτησε η διαπραγμάτευση. Πραγματικά κράτησε πάρα πολύ καιρό. Θα ξεκινήσουμε στις 2 και 4 τη συνεδρίαση της ΕΚΟΝ με τον πρόεδρο του CFTC, τον κύριο Μασάντ. Meeting is closed.